Όσον αφορά ε, τώρα ε, ε, την, ημερησία διάταξη, είπαμε ότι έχουμε αυτό το, το σχέδιο κειμένου της 2 Ιανουαρίου του 2010. Έχετε λάβει αυτό το κείμενο και τώρα θα συζητήσουμε το θέμα στην ημερησία διάταξη. Πρώτον, ξεκινούμε από την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου. Οπότε η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων ενέκρινε την έκθεση του κυρίου Ραπκάε που αφορά την άρση ασυλίας του κυρίου Βίκτορ Ουσπάσκιτς. Πολιτικές ομάδες απεφάσισαν ομόφωνα. Αποφάσισαν η ψήφιση να γίνει αύριο το μεσημέρι θα γίνουν και άλλες ψηφοφορίες. Σας επαναλαμβάνω, πρόκειται για την έκθεση ΡΑΠΚΑΕ που αφορά την ε, άρση ασυλίας του κ. Πάσχης θα γίνει ψήφιση αύριο. Αυτά όσον αφορά την σημερινή ημερησία διάταξη δυνάμει του κανονισμού. Τέτοιε εκθέσεις, ε, τέτοια αιτήματα ε, θα πρέπει να συζητούνται στην αρχή της Συνόδου. Η κυρία Αντζελίλη, ο κύριος Πιτέλα και άλλοι 40 συνάδελφοι υπέβαλαν έτοιμα αναβολής της συζήτησης για την κυρία Σακίνεχ Μοχαμαντή Αστιάνια. Ζητούν να συζητηθεί αντί για την Πέμπτη, σήμερα Δευτέρα. Κυρία Αντζελίλη, παρακαλώ παρουσιάστε την πρότασή σα το έτοιμά σα. Εάν Α, ο κύριο Πιτέλα, έχετε το λόγο. Ήθελα να πω απλώ ότι είπατε πράγματα σύνετα και τα είπατε με μεγάλο κύρος όσον αφορά την νεαρή γυναίκα στα κίνε. Αλλά άλλο είναι τα λόγια που χειροκροτήθηκαν κιόλα. Και άλλο πράγμα είναι μια επίσημη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πράγμα το οποίο πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι η μοίρα ε, τη γυναίκα αυτή εξαρτάται από αποφάσει που θα ληφθούν μέσα στις επόμενες ώρες. Ακούγονται όλο και περισσότερο φωνές που ζητούν να αλλάξει η απόφαση. Αλλά ε, δεν μπορεί από τις φωνές αυτές να λείψει η φωνή με κύρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό θα πρέπει ε, ε επιγόντως να φέρουμε πιο μπροστά τη συζήτηση αυτή που προβλεπόταν για την Πέμπτη και να την κάνουμε σήμερα. Μαουρό, ε, Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάριο Μάουρο θα ήθελα να μιλήσει υπέρ της πρότασης αυτής. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Παίρνω το λόγο ακριβώς με σκοπό να υποστηρίξω το αίτημα αυτό, γνωρίζοντας ότι ε, μια Ευρώπη που πρωταγωνιστεί ε, στην ε, ε, ειρήνη και στον πόλεμο είναι μια Ευρώπη που παρεβαίνει την κατάλληλη χρονική στιγμή. Ε, προσπαθούμε πολλές φορές να θέσουμε τέτοια ζητήματα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά πιστεύω ότι όταν το απαιτούν οι συνθήκες να ε, ενεργούμε ε, Και γι' αυτό ε, συμφωνώ με όλους τους συναδέλφου που υποστηρίζουν αυτό το αίτημα. Ο σας ευχαριστούμε και τώρα. Πέστε μας αν κάποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο κατά αυτού του αιτήματο. Κατά. Ε, Κυρίε και κύριοι, τώρα θα ψηφίσουμε με αυτές τις προτάσεις. Συγγνώμη, θα ήθελα να παρακαλέσω το δυνατόν γοργότερα να ψηφίσουμε για το κείμενο. Και δεν έχει νόημα σήμερα να συζητήσουμε, αλλά να ψηφίσουμε πολύ υστερότερα. Αυτό ήθελα να πω. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Okay. Καλώ λέει ο πρόεδρο, οπότε ψηφίζουμε. Ποιοι είναι οι υπέρ τη πρόταση Αντζελίλη και Επιτέλα να συζητηθεί σήμερα το θέμα. Ποιοι είναι κατά, ευχαριστούμε, αποχές, άρα εγκρίνεται η πρόταση. Επομένως, έχουμε τώρα την ε, συζήτηση αυτήν η οποία θα τελεστεί σήμερα. Το πρώτο θέμα της ε, ολομελίας όταν ολοκληρωθεί η έγκριση της σημερινής διατάξεως. Στις 7 η ώρα μια προθεσμία για υποβολή διαφόρων προτάσεων ε, για, κάποιες, ε, για κάποια ψηφίσματα και για τα κοινά ψηφίσματα, τα υπόλοιπα, αύριο το μεσημέρι. Αυτές είναι οι πρώτες προθεσμίες που εκπνέουν. Στις, ε, μέχρι τις 7 η ώρα θα πρέπει να υποβάλλεται τυχόν προτάσεις για ψηφίσματα. Και Παναλαμβάνει ο πρόεδρος άλλη προθεσμία, η εκπνέει αύριο το μεσημέρι για τα κοινά συνήθη ψηφίσματα. Οι ψηφοφορίες θα γίνουν το μεσημέρι της Τετάρτης. Τότε θα ληφθεί απόφαση με την ε, ε, ψηφοφορία. Αυτή είναι η ταχεία διαδικασία για την συγκεκριμένη ε, συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε τίποτα άλλο για τη σημερινή ημερησία διάταξη. Δεν βλέπω κανείς να ζητεί το λόγο, ούτε έχουν υποβληθεί προτάσεις για Τρίτη ή Τετάρτη. Όμως θα γίνει συζήτηση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο. θα ήθελα ένα λεπτάκι να δούμε το εξής. Η συγκεκριμένη συζητηση είναι πάρα πολύ σοβαρή και η οποία για πρώτη φορά διεξάγεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα θέλαμε να προσέξουμε σε αυτή την συζήτηση τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο υποδεικνύει την κατεύθυνση που θα πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει όλους μας γιατί θέλουμε τέτοιου είδου ε, εικόνα να προβληθεί για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια εικόνα ευθύνη και υπευθυνότητα είναι και το θέμα τη καινούργια συνθήκη στην Ήτλη Λισαβόνα που μα ε, προσδίδει περισσότερε αρμοδιότητε, Πολύ σοβαρά πρέπει να πάρουμε μέρο στη συγκεκριμένη συζήτηση που θα γίνει. Όπω δεν γνωρίζετε, η διάσκεψη των Προέδρων ήδη την Πέμπτη συνεζήτησε το θέμα, οπότε και μιλήσαμε για το πόσο λίγοι βουλευτέ προσέχουν να συζητήσουν σε κάποια θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Πολύ, πολύ λίγοι. Ιδίω όταν συζητάμε θέματα ε, θεσμικά και διαθεσμικά. Σε αυτή τη διάσκεψη των Πρόεδρων πριν από τέσσερις μέρες μιλήσαμε επαναλαμβάνω, για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά κάποιο τρόπο ε, προπαρασκευαστικά. Αύριο στις 9 πρόκειται να γίνει αυτή η συζήτηση εδώ εν ολομελία οι δε επικεφαλής των πολιτικών ομάδων ζήτησαν να συμμετάσχουν όλοι οι βουλευτές σε αυτή τη συζήτηση. Από τον Ιούλιο οι επικεφαλής των ομάδων απεφάσισαν να μην γίνουν την ίδια ώρα άλλες συνεδριάσεις. 9 με 11 και μισή το πρωί. Δεν θα υπάρξει άλλη συνεδρίαση, δεν θα γίνει άλλη συζήτηση, άλλο, άλλη, άλλη εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, που να ανταγωνίζει το ΣΥΠΗΝ τη ζήτηση αυτή που θα κάνουμε εδώ. Και επίση αποφασίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων ότι θα υπάρξει ειδικό έλεγχος ποιοι παρίστανται και ποιοι απουσιάζουν από αυτή τη συζήτηση. θα σας ζητηθεί να πατήσετε ε, σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές κατά την συζήτηση ένα κομπάκι. Στις 6.30 απόψε θα συνεδριάσει το Προεδρείο. Εκεί θα προτρέψω τη συζήτηση για το ποια μέτρα θα ληφθούν σχετικά δηλαδή πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για την προσέλευση, την παρουσία των βουλευτών. Ακόμα δεν ξέρουμε τι απόφαση θα ληφθεί, δεν μπορούμε να την προδικάσουμε, όμως προσωπικά παρακαλώ όλοι να έρθετε σε αυτή τη συζήτηση αύριο. Αλλά παρακαλώ να έρθετε και σε όλες τη υπόλοιψη αυτή τη ε, θητεία. Στι 9 θα αρχίσει αυτή η συζήτηση και προσωπικά τον καθένα από εσά τον παρακαλώ να έρθει. Να έρθει γιατί η συζήτηση αυτή είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Είναι πάρα πολύ σημαντική και για την εικόνα που θα δώσει το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να λάβουμε τι ευθύνε μα όσον αφορά το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα δεν έχουμε συζητήσει, δεν έχουμε κρίνει πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες, τα στοιχεία αυτά για το ποιος είναι παρόν κατά την συζήτηση. Αυτά θα το αποφασίσει το Προεδρείο σήμερα. Ε, κολέγα Πόσελτ, νούμερο 749. Πόσελτ, ε, κύριε Πρόεδρε, Είμαστε ελεύθερα εκλεγμένοι βουλευτές και με καθαρή τη συνείδηση θέτουμε προτεραιότητες. Είχα υπόψη να συμμετάσχω στη συζήτηση αύριο και το εξετάζω αυτό πάλι εκ νέου, αλλά το λέω με σαφήνεια αν έχουμε οποιοδήποτε είδους ελέγχους ηλεκτρονικούς δεν θα συμμετάσχω και αν άλλα μέτρα καταμέτρησης υιοθετηθούν από την διοίκηση τότε το κτίριο θα το εγκαταλείψω κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Είχα υπόψη να προσέλθω, αλλά αυτές οι μέθοδοι είναι κατά των ελεύθερα εκλεγμένων βουλευτών και είναι αναξιοπρεπείς μέθοδοι. Ευχαριστώ. Dziękuję bardzo e, za wypowiedź. Σας ευχαριστούμε για αυτό το σχόλιο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λάτφορντ. Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Πόσελ. Πιστεύω ότι το τραγικό ε, είναι ότι αν, είχαμε, αν, είχατε απλώς ε, ενθα, αν μας είχατε απλώς ενθαρρύνει να είμαστε παρόντες, σίγουρα θα είχα σεβαστεί το κύριο σας και την ηγεσία σας. Είχα και εγώ την πρόθεση να παραστώ. Αν είμαι όμως ε, παρούσα αύριο το πρωί, σίγουρα δεν θα συμμετέχω στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και νομίζω ότι θίγεται η φήμη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Προέδρου Μπαρόζο. γιατί θα πει ο κόσμος ότι το Προεδρείο κάνει αυτή την πρόταση γιατί διαφορετικά ε, φαίνεται ότι θα φανεί ότι μόνο επειδή μας υποχρεώνεται θα έρθουμε να ακούσουμε τον Παρόζο. Πραγματικά είναι ε, σαν να ε, πυροβολούμε τον εαυτό μας και πραγματικά είμαι κατάπληκτη που το Προεδρείο κάνει αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Απίθυνα έκκληση σε εσά να είσαστε παρόντε κατά τη συζήτηση πολλέ φορέ πιο πριν κιόλα. Και η συζήτηση σίγουρα θα είναι πολύ έντονη. Άσχετα από την απόφαση του Προεδρείου, νομίζω πάρα πολλοί θα είναι παρόντες. Ο κύριος Ντόλ. Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονό ότι στη διάσκεψη των Προέδρων αποφασίσαμε και αισθάνομαι και υπεύθυνο, έστω και δεν ήμουν παρόν προσωπικά, αναλαμβάνω όμω την ευθύνη μου. Ε, αποφασίσαμε τα εξή. Πρώτον, ότι σαν διάσκεψη των Προέδρων προτείνουμε την ε, ε απόφαση που είπατε εσεί ε, στι συνεδριάσει των ομάδων, ε, των πολιτικών ομάδων. Οι πολιτικέ ομάδες όμως, οι δική μου και οι άλλε, δεν συμφώνησαν με την απόφαση που πήραμε στη διάσκεψη των Προέδρων που την πήραμε ίσως και υπερβολικά βιαστικά. Εγώ λοιπόν θα πρότεινα να ε, επανέλθουμε στο Προεδρείο, να αναλύσουμε την πρόταση αυτή μαζί με τους επιφελείς των πολιτικών ομάδων, γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές συζητάμε αλλαγές, αλλά ο μορτίνο ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο το παριστάνουμε. Δεύτερον, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω αγαπητοί συνάδελφοι, πόσες φορές κάναμε τη συζήτηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε μαζί του. Υπάρχουν όμως 27 επίτροποι που έρχονται και κάθονται εδώ ε, ναι, έρχονται συνήθω οι επιτροποί όταν γίνονται οι συζητήσει. Και μιλάει και ο πρόεδρο Μπαρόζο και υπάρχουν εδώ και οι υπεύθυνοι, οι επικεφαλεί των πολιτικών ομάδων και η αίθουσα είναι άδεια. Γι' αυτό υποστηρίζω ε, την πρόταση αυτή. Να μην εφαρμόσουμε αυτό που σκεφτήκαμε στη διάσκεψη των Προέδρων, να το ξαναδούμε, να το ξαναζητήσουμε στις πολιτικές ομάδες και να εφαρμόσουμε την παλιά μέθοδο, αλλά να ζητήσουμε από όλα τα μέλη να δείξουν ε, υπευθυνότητα και να ε, παραβρεθούν στην πολύ σημαντική συζήτηση που θα κάνουμε εδώ αύριο το πρωί για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ και ζητώ να γίνει μια συνετή ανάλυση στο Προεδρείο ίσως ε, πιο συνετοί από αυτοί που κάνουν οι πρόεδροι των πολιτικών, οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων και να συνεχιστεί αυτή η δημοκρατική συζήτηση σαν ε, συζήτηση μεταξύ υπεύθυνων ανθρώπων. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι το προανέφερα ότι το Προεδρείο θα συζητήσει αυτό το θέμα σε μια ώρα περίπου από τώρα. Είμαι πεισμένος ότι το Προεδρείο θα εξετάσει τα υπέρ και τα κατά ως επιχειρήματα και θα λάβει υπόψη όλα τα σχόλιά σας τα οποία έχουν εκφραστεί και εδώ επίσης. Φυσικά δεν υπάρχει κάποια αναφορά στον εσωτερικό μας κανονισμό για αυτό. Δεν θα ήθελα να χρονοτριβούμε τώρα και να μακρηγορούμε με αυτή τη συζήτηση. Με ιδιαίτερη σοβαρότητα αντιμετωπίζω το θέμα και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά απόψε θα υπάρξει μια άλλη διάσκεψη πρόεδρων μετά από τρεις μέρες την Πέμπτη. Παρακαλώ λοιπόν αφήστε τα αρμόδια σώματα να αναλύσουν το ζήτημα και θα ληφθεί απόφαση από το Προεδρείο απόψε. Θα ήθελα λοιπόν να μην προβείτε στο να κάνετε σχόλια τώρα. Γνωρίζω τις ενστάσεις και αντιρρήσεις σας. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω να σταματήσουμε τώρα αυτή τη συζήτηση εδώ και τώρα. Όλοι έχουμε ακούσει τα συγχαρητήρια μετά το πρώτο σχόλιο εναντίον αυτής της πρότασης σε αυτό το ζήτημα. Και τώρα γνωρίζουμε τις ενστάσεις ε, που έχουν διατυπωθεί. Θα ήθελα να ολοκληρωθεί τώρα, να τερματιστεί αυτή η συζήτηση και πάλι με επανάληψη της έκκλησης να είσαστε παρόντες αύριο στις 9 στην Ολομέλεια. Θέλουμε να είναι μια πανηγυρική, σοβαρή συζήτηση στην Ολομέλεια. Θα θέλαμε με κάθε σοβαρότητα να δείξουμε την ευθύνη και ότι είμαστε υπεύθυνοι. Και θα υποβάλουμε, θα δείξουμε την εικόνα του Κοινοβουλίου. Θα δώσουμε με κύρος την εικόνα του Κοινοβουλίου, ανταποκρινόμενοι στον ρόλο μας, όπως θέλουμε να μας βλέπουν. Θα συζητήσουμε λοιπόν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνω έκκληση να είσαστε λοιπόν παρόντες εις εννέα στην Ολομέλεια εδώ σε αυτή την αίθουσα. Εντάξει. Και στην συνέχεια ένα μόνο σχόλιο υπάρχει για την Πέμπτη. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας που ελήφθη πριν από ένα λεπτό, αυτό που θα κάνουμε είναι θα επισπεύσουμε αυτή τη συζήτηση για την κυρία Σακίνη Νταστιάνη. Θα διεξαχθεί αυτή η συζήτηση λοιπόν άμεσα με αυτές λοιπόν τις αλλαγές η ημερήσια διάταξη υιοθετείται. Ο κύριος Περόνι. Πρόεδρε, δεν θέλω να ξανανοίξω τη συζήτηση για τον έλεγχο των παρουσιών αύριο, αλλά και μετά την παρέμβαση του συναδέλφου Τόλ, εφόσον στο Εφόσον η ατζέντα, η ημερήσια διάταξη μπορεί να τοποποιείται από την ημερήσια διάταξη, ζητάω να ψηφίσουμε εδώ για την απόφαση της διάσκεψης των Πρόεδρων, να ψηφίσουμε εδώ για την απόφαση αυτή, με σκοπό ενδεχομένως να την τροποποιήσουμε. Μπορούμε. Μπορούμε να ψηφίσουμε από αυτού αύριο. Αυτό που θα ήθελα είναι να αναμείνουμε να ληφθεί πρώτα η απόφαση του Προεδρείου. Εντάξει. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την πρώτη μας συζήτηση επί του πρώτου θέματος ε, απόψε. Αυτό που θα κάνουμε είναι θα ακούσουμε τον εισηγητή πρώτα. What we should, the, the first point is, is the first. Yeah.